Επαναλαμβάνεται η συνεδρίαση, τα πρακτικά τη χθεσινής συνεδρίασης και τα κείμενα τα οποία έχουν εγκεκριθεί, έχουν δημοσιευθεί, υπάρχουν αντιρρήσει σχετικά. Εάν όχι, θεωρούνται ότι έχουν εγκριθεί τα πρακτικά.